az ennek Good afternoon, ladies and gentlemen. Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι. Παρότι καθυστερήσαμε με το τέλος των ψηφοφοριών, Πρέπει να συνεχιστούν οι εργασίες μας και πρέπει έτσι να συνεχίσουμε. Θα συνεχίσω στα Ουγγρικά, στη γλώσσα μου. Μάλιστα, λοιπόν, Α, ε, τα πρακτικά της χθεσινής συνεδρίασης είναι στη διάθεσή σας. Υπάρχουν κάποια σχόλια, κάποιες αντιρρήσεις, ενστάσεις. Δεν υπάρχουν. Έτσι λοιπόν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι εγκρίνονται τα πρακτικά της ε, χθεσινής